Λοιπόν, παρακαλώ καθίστε στις θέσεις σας. Liebe Kollegen, bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Ich möchte Ihnen... Θα ήθελα να σας κάνω δύο ανακοινώσεις εισαγωγικά. Πρώτον, τα πρακτικά της συνεδρίας των συντονιστών σας έχουν υποβληθεί. Είναι μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, όποτε και αν τελειώσει σήμερα, αύριο δεν έχουν υποβληθεί τροπολογίε, θα θεωρηθεί ότι εγκρίνουν τα πρακτικά αυτά συνεδρίες των γνωστών. Δεύτερη παρατήρηση. Οι συντονιστέ στη συνεδρίασή του σήμερα συμφώνησαν να ψηφίσουμε κάθε τροπολογία μόνο ηλεκτρονικά. Έχουμε 850 ψηφοφορίες περίπου. Χρειάζεται πάρα πολλής χρόνος. Θα αρχίσουμε λοιπόν έτσι και θα δούμε μετά από μία ώρα, θα ελέγξουμε εάν έχουμε πιθανότητες να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Εάν δεν τα καταφέρουμε σήμερα, έχουμε προβλέψει συνεδρίαση αύριο, θα πρέπει να συνεχίσουμε αύριο. Αν τα καταφέρουμε, θα μπορέσουμε αύριο να μην χρειαστεί να συνεδριάσουμε. Θα σας το πω, θα σας το πω, είναι ευθέτω χρόνο. Ε, δεν μπορώ να σας πω τώρα τίποτα. Πρέπει να κάνω κάποιες ανισώσεις, συνάδελφε Κασπαρή. Εάν μπορούμε να προχωρήσουμε ηλεκτρονικά, σας λέω ψηφίστε τώρα και τέλος. Δεν θα, δεν θα ρωτάω ψήφισαν όλοι και λοιπά. Ναι, μπορούμε κάπως να επιταχύνουμε τη διαδικασία. Εντάξει. Τρίτη παρατήρηση. Έχουμε web streaming. Καταγράφεστε όλοι λοιπόν. Θέλουμε να, κάνουμε, να δώσουμε μια καλή εντύπωση προς τα έξω, να είσαστε φιλικοί προς αλλήλους και προς εμέ, δεν θέλουμε να τσακωθούμε, προβλήματα υποχρεωτικά. Παρακαλώ, είναι όλοι στις θέσεις τους εκείνοι που θέλουν να ψηφίσουνε. Θα κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία για να μην είναι υπερβολικά πολλοί οι ψηφίζοντες. Λοιπόν, ψηφίζουμε τώρα, δοκιμαστικά. Also es geht nur elektronisch. Μόνο ηλεκτρονικά, μόνο ηλεκτρονικά. Όποιος δεν έχει την κάρτα μαζί του δεν μπορεί να συμμετάσχει στην ψηφοφορία. Πολύ απλό. Θα μα πει ο Αλμπέρτο τι γίνεται. 24 συμμετείχαν στην ψηφοφορία μέχρι στιγμή. Πέρασε η ε, ψηφοφορία. Also, ich wiederhole nochmal von der PPE 14. ΕΛΚ 14. Μπορώ να συμμετάσχω στην ψηφοφορία. Για να ψηφίσουν όλα τα μέλη του ΕΛΚ. Μόνο το ΕΛΚ παρακαλώ. Μόνο το ΕΛΚ να δούμε πώς είναι. Als abstimmungsberechtigt bis jetzt sind 13 anwesend. 13 είναι παρόντος. Ένας μπορεί ακόμα να προσθεθεί. Ωραία. Α, η αντιπρόεδρος μου εδώ. Εντάξει, ωραία. Όλα τα μέλη των σοσιαλιστών παρακαλώ. Εννέα μπορούν να είναι. Σοσιαλιστές, μόνο οι σοσιαλιστές. Εννέα, εντάξει οι άλλοι δεν είναι τόσο πολύ τους βλέπω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, μπορούμε να αρχίσουμε τώρα τις ψηφοφορίες. Λοιπόν, εάν ψηφίζει κανεί παραπάνω θα το δούμε και θα σας το πούμε. Ωραία. Άρχονται λοιπόν οι ψηφοφορίες. Σημείο προφορική ερώτηση για την έκθεση David Martin για τη με το ΚΑΡΙ Φόρουμ. Εισαγωγικά σας κάνω και άλλη μια ανακοίνωση. Ξέρετε, ότι έχουμε δυναμωμένη συνεργασία με την Επιτροπή ΤΕΒΕ. Ξέρετε και τη σχετική απόφαση που ελήφθη στην ΑΦΚΟ. Ανεξάρτητα από αυτό, Έχουμε συμπεριλάβει σε αυτό το φάκελο εκείνα τα σημεία της Επιτροπής Ανάπτυξης που δεν ψηφίζουμε γιατί είναι δική τους αρμοδιότητα. Και θα ήθελα να σας ενημερώσω, να σας ενημερώσω λέω, ότι η Επιτροπή ΔΕΔΕ όσον αφορά το ΒΓ ΔΕΛΤΑ όσον αφορά μία σειρά τροπολογιών έχει αναφέρει θετικά όπως το 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 21. Για ενημέρωσή σας μόνο. Και περνάμε τώρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Sorry. Uh, I'm very happy for the developments. Χαίρομαι για την άποψη της Επιτροπής Ανάπτυξης. Αν νομίζω ενισχυμένη συνεργασία όχι για το ψήφισμα. We don't have enhanced cooperation on the resolutions. Για τη σύμφωνη γνώμη, όχι για το ψήφισμα. Εκεί είναι η σημαίνει συνεργασία. Πρόεδρος. Η απόφαση που ελήφθη προηγουμένω είναι ότι θα υπάρχει ενδυναμωμένη συνεργασία μεταξύ των δύο επιτροπών υπό την ηγεσία της ΣΥΝΤΑ. Το κάναμε αυτό. Εκεί προσανατολιστήκαμε. και είπαμε ότι ορισμένες ε, έχουν ψηφιστεί από εκείνους, ε, ορισμένες εγώ σας ενημέρωσα απλώς. Νομικά δεν έχει καμία, καμία, ξέρει, γι' αυτό σας το είπε έτσι. Γενικά. Also, weil die... Γιατί τότε στην απόφαση της Διάσης του Προέδρου είχε ληχθεί ότι και οι δύο επιτροπές από κοινού θα πρέπει να προετοιμάσουν αυτό το ψήφισμα. Γι' αυτό ακολουθούμε αυτή τη διαδικασία. Ελπίζω να απάντησα στο ερώτημά σα. Τα άλλα ήταν ε, απλώ μια ενημέρωση τέβε. Δεν χρειάζεται να το λάβετε υπόψη, σα το είπα απλώ για ενημέρωσή σα. Λοιπόν, εμεί ψηφίζουμε τώρα το δικό ψήφισμα. Ωραία. Σχέδιο προφορική ερώτηση. Συμβαστική τροπολογία 1. Ψηφίζουμε που έχετε πλήρως εκεί. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Ένας σοσιαλιστής θα πρέπει να αποσύρει την κάρτα του. Είναι ένας παραπάνω εδώ. Προφορική ερώτηση ψηφίζουμε. Επαναλαμβάνω. Σας παρακαλώ συνάδελφοι, σας παρακαλώ. Έχουμε 850 ψηφορίες μπροστά μας. Ακούστε τον πρόεδρό σας. Μπορεί να υπάρξουν και σφάλματα στη δικασία ψηφοφορίας, αλλά είπα ξεκάθαρα ότι θα ψηφίσουμε το σχέδιο προφορικής ερώτησης. Συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 1. Την έχετε ενώπιόν σας. Είναι προσαρτημένη στο τέλος. Αυτό ψηφίζουμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, στην πρώτη σελίδα. Κύριε Αντιπρόεδρε, σας παρακαλώ, μην μιλάτε όλοι ανακατεμένα. Για τρίτη φορά σας το λέω, έχετε και στο συντονιστή σας. Ψηφίζουμε τώρα το σχέδιο προφορικής ερώτησης. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. 17 υπέρ, 10 κατά. Εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε τις τροπολογίες για το σχέδιο ψηφίσματος. Είδατε, είδατε. Ξέχασα. Πρέπει να ψηφίσουμε το σύνολο της Προφορική ερώτηση. Όλες οι άλλες έχουν αποσυρθεί. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα κατά βάση, αλλά πρέπει για να είμαστε εντάξει να ξαναψηφίσουμε το σύνολο της, του σχεδίου προφορικής ερώτησης. Άρχιτη ψηφοφορία. Το ΕΛΚ έχει έναν ψηφίσοντα περισσότερο. Ωραία τώρα. Λοιπόν, τη ψηφοφορία. 23 υπέρ και 2 απόχέ. Ε, συγχαρητήρια, Ντέβιτ, έγινε δεκτό αυτό. Περνάμε τώρα στι τροπολογίες για το σχέδιο ψηφίσματος. Συμβαστική τροπολογία παριθμών 1, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορία. 25 εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. 12 υπέρ 13 κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 18. Άρχισε ψηφοφορία. Πέρας. Δύο ψήφοι υπέρ 18 κατά 5 αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 21. Άρχισε ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 23. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 24 άρχιδη ψηφοφορία. Το ΑΕΛΚ έχει ένα παραπάνω. Εντάξει τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. 14 προς 14. Απορρίπτεται. Τροπολογία 26. Άρχιδη ψηφοφορία. Πέρας. Ε, 12 προς 16. Τροπολογία 30. η ψηφοφορια ψηφοφορία. Πέρας. 17-11 εγκρίνεται. Τροπολογία 31. η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. Τροπολογία 32. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία υπαριθμών 1. Διαφωνεί κανένα με την προφορική τροπολογία? Όχι. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 33. Άρχιε ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Ο κατάλογο προφορά που έχω δεν είναι πολύ επίκαιρο. Λυπούμε. Δεν υπάρχει κατασμήντα ψηφορία, μου λέει η γραμματεία. Also, mich nach der Λοιπόν, εγώ ακολουθώ τον κατάλογο ψηφορία που μου έχει προετοιμάσει η γραμματεία. Δεν υπάρχει κατασμήντα ψηφορία. ό,τι και αν θεωρούν οι πολιτικές ομάδες πρέπει. Εδώ δεν υπάρχει κατευθυνότητα ψηφοφορία. Άρα. Ευχαριστώ. Ζητήσαμε χωριστή ψηφοφορία. Δεν ξέρω τι ακριβώ έγινε. Το έχουμε στα εγγραφά μα αυτό. Χωριστή ψηφοφορία. Το ζητήσαμε. Εδώ και κάμποσο καιρό. Δεν ξέρω τι συνέβη. Η γραμματεία το ξέρει. Η Γραμματεία το ζήτησε. Δεν υπάρχει ούτε τώρα ψηφίσαμε κατά οπότε. Ωραία. Μου λέει μόλις τώρα η Γραμματεία ότι υπευλήθη καθυστερημένα το έτοιμά σα αυτό. Αυτό ο κατάλογο που έχει τη γραμματεία που είναι δεσμευτικό δεν χρειάζεται κατά την ψηφοφορία. Α προχωρήσουμε πάντω. Το πατρίσμα έδωσε λύση. Προχωράμε στην απολογία 23 λέει ο πρόεδρος. Άρχη ψηφοφορία. Α, 34 εννοούσα. Ναι, ναι, ναι, ναι. 34. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 35. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 36. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρο... Απορία όσο πάει και πιο πολύ. Τροπολογία 37. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 38. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 39. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Θα μπορούσαμε να το ψηφίσουμε όλα αυτά μαζί. Τροπολογία 40. Άρχεται. Πέρας πληροφορίες. Εγκρίνεται. Γιατί 41 θέλουμε αν γίνεται χωριστή ψηφοφορία. τονίζει τους κινδύνους που η εγκατάλειψη εθνικών πόρων να δημιουργήσει σε αναδυόμενες οικονομίες ενθαρρύνοντας πράξεις διαφθοράς και κακοδιαχείρισης ως προς το εισόδημα. Εκεί, εκεί να γίνει ο χωρισμός, ο διαχωρισμός. Κρίστοφερ, συμφωνείς αυτό ζήτησες και εσύ. Α, συγγνώμη, το 41 σαν ε, σημάνει το μεγάλη διαφορά μεταξύ των δαπανών στις ε, γεωρικές δαπάνες και οικονομική και τεχνική υποστήριξη. Εκεί να γίνει, να είναι η διαχωριστική γραμμή. Θα σας κάνω μια πρόταση. Στον κατάλογο μου δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Γι' αυτό λοιπόν η... θα δείξω πολύ ενοχή. Θα πω, θα θεωρήσω ότι αυτό είναι μια προφορική τροπολογία. Έχει κάποιος κάτι κατά της προφορικής τροπολογίας? Όχι. Θα ψηφίσουμε λοιπόν έτσι σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα της τροπολογίας. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 42. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 43. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 44. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία Συμβιβαστική παρελθόν 2. Άρχισε φορέα. Α, όχι. Πρώτα DV3. TV3, ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 2. Άρχιδη ψηφοφορία εγκρίνεται. Συμβασική τροπολογία παριθμών 3. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 50 καταπίπτει. 54. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απερίπτωτα. 55. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 56. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 57. Άρχιτη ευφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 58. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Ναι, Ρόμπερτ. Το ΕΛΚ αποφάσισε να ψηφίσει υπέρ, όπως και τη συμβαστική 7. Το λεφτό για τους συναδέλφους. Έχουμε συμφωνήσει με το 5 και το 7 με τον David Martin. θα είμαστε υπέρ του 5 και του 7. Θαυμάσια. Θα ψηφίσουμε παρόλα αυτά. Συμβαστική παριθμό 5 άρχεται. Πέρας. Ναι, το βλέπουμε από το αποτέλεσμα. Καταπίπτει 61. Περνάμε στη συμβαστική 6. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 64. <coughs> Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 67. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 68. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 69 άρχεται πέρας απορρίπτεται 7 συμβαστική 7 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται τροπολογία 73 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Απορρίπτεται. 74. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. που 75. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 76. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 8. Άρχισε φορεία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 77. Άρχισε ψηφοφορία. Τροπολογία 80. Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. 81. Άγιο ψηφοφορία. Το ΕΛΚ έχει ένα ψηφίσοντα περισσότερο από ό,τι πρέπει. Πέρασε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. TV4. Άρχιτη ψηφοφορία. περασε Πέρασε. Απορρίπτεται. TV5. Άρχιτη ψηφοφορία. Ich bitte eine Karte rausnehmen. Beendet. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 82. Άρχη ψηφοφορία. Beendet. κρίνεται. Τώρα Τροπολογία 83. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 10. Άρχιε ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 84. Άρχη ψηφοφορία. Πάλι έχει το έλκανα παραπάνω. Πέρας. Εγκρίνεται. Μου το λέει εδώ το εγγραφό μου, Ρόμπερτ, ότι υπάρχει ένα στο ΕΛΚ παραπάνω. Και όταν μου το δείχνει εδώ πέρα, το λέω. Δεν ξέρω ποιος. Αυτό Αυτόματο γίνεται αυτός ο έλεγχος. Κύριε Αντεπρόεδρο, εδώ μπορεί να το δει και εκείνη ότι δεν είναι δική μου έμπνευση. Το συμβαστική τροπολογία 11 άρχεται ψηφοφορία. Also nochmal den Änderungsantrag 84. Τροπολογία 84 ξανά. Νομίζω ότι ψηφίσαμε. 84 ξανά η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 11. 11, 11. ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 87 και 88 ταυτόσιμες. Άχι ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 90 και 91. Άρχισε ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία. Για την παράγραφο 20. Διαφωνεί κανένας? Όχι. Ψηφίζουμε. Άρχιε ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 92. Δεν φωνεί κανένα. Να ψηφίσουμε ο μπλοκ 92-97. Όχι. Λοιπόν, ψηφίζουμε όλες αυτές. 92-97. Όχι. Ωραία. 92. Άρχισε ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 93. Άγιο ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 94. Άρχισε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 95. Άρχιψη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 96. Άρχισε ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 97. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 98 και 99 έχει την ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 12. Άρχιδη ψηφοφορία. Πέρας. 14 από 14. Απορρίπτεται. Τροπολογία 100. Όχι. Άχι ψεφούρε λέει ο πρόεδρος. Ist ja an. 17 προς 10. Εγκρίνεται. Η ΤΕΒ1 καταπέφτει. Σε δείχνουν προς τα γραμματεία, γιατί το λέει αυτό. Ναι, καταπίπτει. Και 104 έχει αποσυρθεί. 105. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Μητρολογική σκέψη Α. Άρχισε ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Άρχισε ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τρία. Τροπολογία 3. Άρχισε ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τέσσερα. Άρχισε ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η πέντε καταπίπτει. Έξι. Έχει ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 7 κατά 5, 8. Έχει ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 9. Έχει ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 10. Άχι ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 11. Άρχεται. Πέρας εγκρίνεται. Συνδεστική τροπολογία 9. Άρχιδη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Και φτάνουμε στην ψηφοφορία την τελική. Έρικα, εσύ το λόγο. Δύο λεπτά να μας δώσετε για να αξιολογήσουμε την κατάσταση που συμμετείχε. Δύο λεπτά. Ναι, λέει ο πρόεδρος, ναι. Κάθε ομάδα μπορεί να το ζητήσει βέβαια. E λοιπόν, συνονίθηκε με τους αριστές μεταξύ τους. Ωραία. Ερχόμαστε. Τελική ψηφοφορία. Έναρξη. Die Abstimmung ist Πέρας. 17 υπέρ 18, 12 καθά, ε, καμία αποχή εγκρίνεται επί 29 συνολικός ψηφισάντων. Συγχαρητήρια, Ντέβιντ. Ελπίζω να είσαι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα αυτό. Και έτσι μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία, στο, στη συμφωνία. Για τη σύμφωνη, για τη σύμφωνη γνώμη. Μία ψηφοφορία είναι. Άρχιε ψηφοφορία. Πέρας. 15 υπέρ, 13 κατά. Εγκρίνεται. Και μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 16 της ημερησίας διάταξης που αφορά ενδιάμεση φωνή οικονομική εταιρική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Κοινότητα και Ζακτή του Αλεφαντεστού. Σα θέτω το ερώτημα. Χρειαστήκαμε περίπου τρία τέταρτα για το προηγούμενο θέμα. Μονίμως πάγια θα κάνουμε το ίδιο. Θέλετε έτσι. Ωραία, εντάξει. Προφορική ερώτηση. Oral question. Της τροπολογίας όλη η ομάδας. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. Αν πατάτε το κουμπί πιο γρήγορα θα πάμε πιο γρήγορα. Εγώ πρέπει περιμένω όλοι να πατήσουν το κουμπί. Τροπολογία 2, έναρξη. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Εντάξει. Πέρας. Απορρίπτεται. 10. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 11. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 12 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 13. Έναρξη. Και πέρας. Απορρίπτεται. 14. Έναρξη. και πέρασε. Απορρίπτεται. 15. Έναρξη. Πέρασε. Εγκρίνεται. 16. Έναρξη. Πέρασε. Απορρίπτεται. 17. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Έναρξη. Πέρασε. Εγκρίνεται. Με 17 υπέρ, καμία ψήφο κατά και δέκα αποχές. Τροπολογίες στο σχέδιο ψηφίσματος. Σε μπλοκ. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Έναρξη. Εγκρίνεται. δέκα καταπίπτει. δώδεκα σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Ε, έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 1. Ενάρξη. Πέρας. Απορρίπτεται μικρή διαφορά. 19 ένοξη πέρας απορρίπτεται. Και πρόεδρε, νομίζω και διορθώστε με, συμφωνήσαμε ότι για προφορική τροπολογία της συμβαστική 2 συμφωνήσαμε θεωρεί σημαντική την εφαρμογή να αποκατασταθεί ένα δέον εποπτικό σύστημα που να συντονίζεται από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή στην οποία να παίρνουν μέρο μέλη τη Επιτροπής για το Διεθνέ Συμπόριο Επιτροπή Ανάπτυξη, επαρκή ισορροπία για τη διατήρηση του ρόλου στην Επιτροπή για το εμπόριο. Η Επιτροπή αυτή θα πρέπει να λειτουργεί με ευέλικτο τρόπο, συντονιζόμενη με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ένωση ACP, ΑΚΕ, και η εποπτεία αυτή θα πρέπει να ισχύσει μετά την έγκριση της συμφωνίας. Πρόεδρος, είμαστε στη συμβαστική 2. Αυτό που λέτε αφορά την συμβαστική 6 νομίζω. Είναι λίγο νωρίς. Ψηφίσουμε τη 2 και όταν θα έχουμε στην 6 θα γίνει αυτό που προτείνεται. Μία σύντομη διακοπή γιατί έχουμε εδώ επισκέπτες Έχω μία αντιπροσωπεία από το Κοινοβούλιο της Ουγκάντα με τον αντιπρόεδρο της Βουλής Ρεμπέκα Καντάκα. Χαιρόμαστε για την παρουσία σας. Τώρα ψηφίζουμε ένα θέμα που ίσως σας ενδιαφέρει. Τώρα είναι για το ελεφαντοστού και μετά είναι με την Δυτικοαφρικανική Ένωση Κεντρικής Αφρικής στην οποία νίκη η Ουγγάνα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε παρόντες και παρούσες στο Ευρωκοινοβούλιο. Συμβαστική 2. Έναρξη. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25. Έναρξη. Και πέρας. Απορρίπτεται. 26. Έναρξη. Και πέρας. Απορρίπτεται. 28. Έναρξη. Και πέρας. Απορρίπτεται. 29. Έναρξη. Και πέρας. Απορρίπτεται η 30 σε δύο τμήματα. Πρώτο. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. 31. Πέρας. Απορρίπτεται. Την 32. Πέρας. Εγκρίνεται. 33 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 34 ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 35 ψηφίσμα. Πέρασε. Εγκρίνεται. 36 ψηφίσμα. Πέρασε. Εγκρίνεται. Προφορική. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 39. Υπέρ. Ε, ε, έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 40. Καταπίπτει. Συμβαστική 3. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 44. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 45. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Προφορική 1. Αντιρρήσεις. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 46. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίφθηκε. Συμβαστική 5. Ψηφίζουμε. Πέρας. 13-13 απορρίπτεται. 52. Έναρξη. Η 51 ήταν με τον μπλοκ που ψηφίσαμε. Την 52 ψηφίσαμε τώρα. Πέρασε. Εγκρίνεται. Έρικα. Κοιτάξτε, μια που κατέπεσε η συμβαστική 5, η 51 είναι προς ψήφιση ακόμα. Κοιτάξτε, σε μένα στο κατάλογο της ψηφοφορίας λέει κατλείπεται από την ψηφοφορία on block. Και στην αρχή ψηφίσαμε on block. Η πρώτη ψηφοφορία ήταν αυτή. Και γι' αυτό θα ξαναψηφίσουμε τώρα. Εντάξει. Α, ναι, ναι, ναι εγώ φταίω. Εγώ φταίω, λέει κύριε Μαν. 54 έναρξη πέρασε εγκρίθηκε χωριστή ψηφοφορία στην 59 πρώτο τμήμα έναρξη πέρασε απορρίπτεται δεύτερο τμήμα έναρξη Πέρασε. Απορρίπτεται. 60. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 61. Υπέρ. Ε, ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 62 ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. 64 ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. 56 ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. 66 ηλεκτρονικά. Πέρασε. Απορρίπτεται. 69 ηλεκτρονικά. Πέρασε. Απορρίπτεται. 70 έναρξη. Πέρασε. Εγκρίνεται. 73 ηλεκτρονικά. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβασική 4 ηλεκτρονικά. Πέρασε. Εβδομήντα πέντε. ηλεκτρονικά. Πέρασε. Εγκρίνεται. Εβδομήντα έξι. ηλεκτρονικά. Πέρασε εγκρίνεται 78 ηλεκτρονικά πέρας απορρίπτεται Συμβιβαστική 6 με την προφορική τροπολογία που πρότεινε ο Ρόμπερτ. Αντιρρήσεις. Όχι. Το ψηφίσουμε όπως μας εξηγήθηκε πριν. Ηλεκτρονικά. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Ογδόντα ηλεκτρονικά. Πέρασε. Απορρίπτεται. 87 ηλεκτρονικά. Πέρασε. Εγκρίθηκε. 88 ηλεκτρονικά. Πέρασε. Απορρίπτεται την 89 πέρας απορρίπτεται την 90 πέρας απορρίπτεται αιτιολογικές σκέψεις παριθμόν 1 ηλεκτρονικά. Πέρασε. Εγκρίθηκε. δύο καταπίπτει. Τρία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τέσσερα. Πέρας. Εγκρίθηκε. Η 6. Πέρας. Εγκρίθηκε. Η 8. Πέρας εγκρίθηκε η 7 Πέρας. Εγκρίθηκε. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά. Και πέρας. Και εγκρίθηκε με 27 ψήφους, 16 υπέρ, 11 κατά. Εγκρίθηκε. Περνάμε στο σημείο 17 της Μελισσίας Διάταξης. Ενδιάμεση Συμφωνία Οικονομικής και Εταιρικής Σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Κράτης και Κεντρικής Αφρικής. Αρχίζουμε με το σχέδιο προφορικής ερώτησης. Συμβιβαστικό κείμενο σύμφωνα με το παράδειγμα υπερτυπών 1. Άρχιτη ψηφοφορία. eröffnet. Geschlossen. Peres. Δεκατρία προς δεκατέσσερα μπορείτε. Τώρα μου επισκεφτεί η γραμματεία στο γεγονό ότι. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ακούστε με παρακαλώ πρώτα. Μια που απορρίφθη ο συμβιβασμός θα έχουμε ίσως πάνω από 27 αράδες στο αρχικό κείμενο και δεν θα γίνει ενδεχομένω αποδεκτό. Σας το λέω. Μου το είπαν αυτό. Μπορεί. Και τότε δεν έχουμε τίποτα στα χέρια μας. Λοιπόν, περνάμε τώρα στο σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Στο σχέδιο ψηφίσματος, συγγνώμη. Συμβαστική υπαριθμό 3. Άχι ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμό 13. Άχι ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 14 προς 13. Α, όχι. Πρέπει κάτι να ευκρινίσω με τη γραμματεία ένα λεπτό. But nevertheless, maybe we have to do the final vote. The final vote, if you want. Um Με συγχωρείτε πολύ. Μου διέφυγε. Παρακαλώ να επανέλθουμε στο σχέδιο προφορικής ερώτησης για να έχουμε την τελική ψηφοφορία για την τροποποιημένη προφορική ερώτηση. Το ξέχασα αυτό. Άρχισε ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε λοιπόν τώρα στη συνέχεια. Τροπολογία 15. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 17. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 18. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Προφορική παριθμόν 1. Διαφωνεί κανένα κατά τη προφορική παριθμόν 1. Παρακαλώ. Μία αντίρρηση κύριε Πρόεδρε για αυτή την προφορική τροπολογία η οποία είναι νέα παράγραφος και καλύπτεται αλλού και δεν τη λάβαμε και έγκαιρα. Λοιπόν, ξέρετε ότι άμα υπάρχει διαφωνία για προφορική τροπολογία δεν μπορούμε να ψηφίσουμε από αυτόν. Περνάμε στη 19. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 21. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 23. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 24. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολή 25 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Άρχιε ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχιε ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 27. 26, συγγνώμη. Άρχεται η ψηφοφορία. 26. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 27 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με πολύ μικρή διαφορά. Τροπολογία 28. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 29. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 30. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 31. Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία νόη. 9. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 35. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 36. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 37. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 38. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5. Άρχισε ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 45. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Μήπως μπορείτε να αντιδράτε λίγο πιο γλυγορά. Για να προχωρήσουμε πιο γλυγορά. 46. Άρχισε ψηφοφορία. Α, συγγνώμη, καταπίπτει. Ναι, ναι, ναι, Καταπίπτει. Σωστά. Γιατί... Πέρασε η 45, οπότε η άλλη καταπίπτει. Η 46. Βασική τροπολογία 7. Άρχισε ψηφοφορία. Geschlossen. Πέρας. Απορρίπτεται. 14 προ 14. Τροπολογία 48. Άρχισε ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. 32. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 51. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 52. άρχη η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. Πέντε τρία καταπίπτει, πέντε τέσσερα καταπίπτει, πέντε πέντε. Πέρας. Απορρίπτεται. 56. Άρχισε ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 57. Άρχισε ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 60. Άρχισε ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 61. Άρχισε ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και περάμε στην προφορική τροπολογία υπαριθμών 2. Διαφωνεί κανείς? Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν. Άρχισε ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 14 προς 14. Τροπολογία 64. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Επίσης 14 προς 14 απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 10. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 68. Άρχιδη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 69. Άρχιδη. Πέρας. Απορρίπτεται. 70. Άρχιδη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Καταπίπτει 71. 72. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 74. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 75. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 76. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 20. Άρχισε ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 78. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 79. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 81. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 14 προς 14. 82. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 2. Η ίδια προφορική τροπολογία εδώ. Διαφωνεί κανένα με αυτή την προφορική τροπολογία. Όχι. Έχω αντίρρηση. Για τον ίδιο λόγο που ανέφερα πριν. Οπότε δεν θα ψηφιστεί η προφορική τροπολογία αυτή. Και περνάμε στη συμβαστική παριθμό 2. Άρχιτη ψηφοφορία. Don't. Nein. Also, liebe Αγαπητοί συνάδελφοι, Κάτερα ζήτησε το λόγο και είπε ότι διαφωνεί με την προφορική τροπολογία. Όταν ένας βουλευτής διαφωνεί με μια προφορική τροπολογία δεν ψηφίζουμε επ' αυτής. Και γι' αυτό περνάμε στη συμβαστική τροπολογία παριθμών 2. Επ' αυτής ψηφίζουμε αυτή τη στιγμή. Άρχιε ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται με μία ψήφο περισσότερη κατά. Παρακαλώ, στον Φασκαλέρο. Συγγνώμη που σας κάνω να χάνουμε ώρα. Αλλά εγώ ψήφισα το συμβιβασμό 2 που λέει ότι συμμετέχουν τα ε, relevant members από τις δύο επιτροπές. Ε, δεν ξέρω αν αυτό το relevant είναι και ο καλύτερος όρος και ο κατάλληλος όρος για ένα κοινοβούλιο. Ίσως τα ισπανικά δεν είναι καλό το κείμενο σας. Τα αγγλικά είναι πιο σαφές, αλλά έτσι και λίγο απερίφθη, οπότε δεν υπάρχει κανένα λόγο να το συζητάμε. Και έτσι περνάμε στην τροπολογία επαριθμών 22. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Απο... Εγκρίνεται. Καταπέφτει η 83 και η 85 και περνάμε στην τροπολογία υπαριθμών 1. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 1. Άρχη ψηφοφορία. φέρεις. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Άρχιτη ψηφοφορία. 6, 7 και 8 ταυτόσημες όλες μαζί. Άρχιτη ψηφοφορία. 6, 7, 8. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία υπαριθμών 3. Διαφωνεί κανένας? Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην Τελική ψηφοφορία. Άρχισε ψηφοφορία. Πέρας. 25 υπέρ, 3 κατά, καμία εποχή. Ωραία. Είναι λοιπόν. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. ε, υπερψήφισε, μπορούμε να του δώσουμε συγχαρητήρια. Και περνάμε τώρα στην Συμφωνία Οικονομική Εταιρική Σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γκάνα. Ψηφίζουμε το σχέδιο προφορική ερώτηση καταρχήν. On Άρχισε η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστικό κείμενο. Σύμφωνα με το παράδειγμα υπ. 1. Άρχισε η ψηφοφορία. Προφορική τροπολογία. Προφορική τροπολογία για το παράθυμα 1. Στο παράθυμα 1 μάλλον. Στην προσπάθεια να δημιουργήσουμε αρμονία και καλοπιστία στην Επιτροπή μας υπέβαλα μια προφορική τροπολογία στο κείμενο του συμβιβασμού. Συνεπώς, αν γίνει δεκτή η προφορική τροπολογία, θα έπρεπε τέλει να ψηφίσει υπέρ. Αλλά καλό το συντάξει να ψηφίσουμε το συμβαστικό κείμενο χωρίς την προφορική, τροπολογία το ΕΛΚ θα ψηφίσει κατά. Δεν ξέρω αν θέλετε να διαβάσω το κείμενο. Μπορώ, αν θέλετε. Δεν ξέρω, είμαι σαφής. Κοιτάξτε, ναι, εγώ δεν είχα το σωστό κατάλογο ψηφοφορία προηγουμένω και γι' αυτό δεν είχα ε, ζητήσει να ψηφιστεί η προφορική τροπολογία. Λοιπόν, περνάμε τώρα στην προφορική τροπολογία που αναφέρεται στο παράδειγμα περιθμών 1. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και έτσι δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε το συμβαστικό κείμενο και περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. κρίθι. Και περνάμε τώρα στο σχέδιο ψηφίσματος. Also ich bin gerne bereit, wir haben es jetzt nach Είναι 4.30, μάλιστα 5 παρα 25. Θέλετε να συνεχίσουμε όπως μέχρι τώρα. Ωραία. Μέχρι 6.30 έχουμε σήμερα και αν δεν προλάβουμε θα συνεχίσουμε αύριο προς 9. Θα δούμε, θα δούμε. Ωραία. Ψηφίζουμε τώρα στο μπλοκ. Το μπλοκ. Άλλη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Το ελέγξαμε αρκετά. Δεν πρόκειται να ελέγξουμε ξανά. Εντάξει, να το υποβάλλετε στην Ολομέλεια και να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια. Ψηφίσαμε. Ψηφίσαμε σωστά. Δεν μπορούμε να ξαναεπανέλθουμε. Λυπούμε. Λυπούμε. Τροπολογία περιθμού 2. Συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 2. Πέρας ψηφοφορίες. Τροπολογία υπαριθμών 92. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παρακαλώ. Πρέπει λίγο να γίνουν πιο σαφή τα πράγματα λοιπόν, και μάλλον εγώ. Ψηφίσαμε το την τελευταία σχέδιο ερώτηση. Ψηφίσαμε. Ψηφίσαμε, ναι, ρε Ναι, ναι, ψηφίσαμε. Ψηφίσαμε. Και περνάμε τώρα. Στη συνέχεια. Τροπολογία 32. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 33. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 34. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 36. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 37. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 39. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Σαράντα. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Σαράντα ένα. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 42. άρθη ψηφοφορία. Πέρες. Απορρίπτεται. 43. Άρχεται. Α, συγγνώμη, ναι. Παράγραφος 5. Σωστά. Παράγραφος 5. Το αρχικό κείμενο της παραγράφου 5. Έχει ζητήσει γνωστή ψηφοφορία από την ομάδα ΕΛΚ ΕΔΕΛΤΑ. Και κατά τμήματα μπορεί να μας το πει αυτό η ομάδα του ΕΛΚ. Πού θέλει κατά τμήματα ψηφοφορία. Στο κατάλογο ψηφοφορία μου λέγεται παράγραφος 5 αρχικό κείμενο Κατά τμήματα ξεχωριστή ψηφοφορία έχει ζητηθεί από την ομάδα ΕΛΚΑ Τι, τι ξεχωριστό. Δεν λέει τίποτα. Α, την παράγραφο εννοείται ξεχωριστά. Α, ωραία, λοιπόν, ψηφίζουμε την παράγραφο 5 αυτή του αρχικού κειμένου, άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Το Τροπολογία 43. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 44. Έχει ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 45. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 49. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 50 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 51 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Και είναι στο μπλοκ, απερίφθη έτσι. 52. 52. Άλλη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 54. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 55. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 56. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 57. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 58. Άρχεται. Πέρες. Απορρίπτεται. 60. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 59. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 61. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 62. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 65. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 66. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6. Άρχεται. Πέρας λέω. Εγκρίνεται. Τροπολογία 70. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 75. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 76. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 77. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 78 άρχεται πέρας απορρίπτεται 79 άρχεται πέρας απορρίπτεται 80 άρχεται Πέρας. Απορρίπτεται. 81. Άρχιδη η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 82. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 83. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 84. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 85. Άρχη ψηφοφορία. Θα το ονειρεύουμε όλη τη νύχτα. Λοιπόν, εγκρίνεται. 86. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 87. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 88. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 90. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 93. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 94. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 95. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 96. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 97. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 98. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 99. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δεν είσαστε ο μόνο που έχει η Κρίσοφερ νομίζω. 101. Άρχη ψηφοφορία. Εκατόν ένα λέω. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 102. Άρχιτη ψηφοφορία. 102. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 103. Άρχινη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 104. Άρχινη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 105. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 107. Άρχεται η ψηφοφορία. Okay, sorry. Okay, yeah. Trying to get some consistency in the report. Για να μην υπάρχουν ανακολουθίες στο κείμενο. Θα κάνω την προφορική τροπολογία που, ε, με την οποία συμφωνεί και ο Ρόμπερτ, αν θυμόσαστε. Αν θέλετε μπορώ να σας την επαναλάβω. Όχι, δεν χρειάζεται να επαναλάβετε. Διαφωνεί κανένα προ την ε, προφορική αυτοπολογία που είχε βάλει προηγουμένω ο Ρόμπερτ. Όχι. Ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροποποιημένη της μορφή. Αλλά πρώτα πρέπει να ψηφίσουμε 107, ε. Βιαστήκατε κάπως, στην Η 107, την 107 ψηφίζουμε πρώτα. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Απεριφθεί. Λοιπόν, περνάμε τώρα στην συμβαστική τροπολογία υπερεθμών 7 Πρέπει να έχω και έναν τρίτο κατά. Ναι, ναι, να είναι ένα το. Συμβαστική τροπολογία 7 με την προφορική τροπολογία. Το είπα, υπό τη μορφή της προφορικής τροπολογίας. Λοιπόν, άρχισε η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και περνάμε στην συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 1. Άρχεται ψηφοφορία. Άρχισε ψηφοφορία λέω. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία παριθμών 3. Άλλη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία παριθμών 4. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 5. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 7. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα παραγγεία παριθμών 8. Έχει ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Μπλοκ. Ψηφίσαμε. Τροπολογία 10. Άχι ψηφοφορία. Δέκα. Ναι, 10, 10, 10, 10. Πέρα Απορρίπτεται. Τροπολογία 15. Άρχισε ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. Σα είπα, τη νύχτα θα, στο όνειρό μου θα λέω άρχεται πέρας, άρχεται πέρας. Λοιπόν, 16 τώρα, άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 18. Άρχιψη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 20. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 23. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 26. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία παριθμών 1. Άρχισε ψηφοφορία. Πέρασε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Και φτάνουμε στη τελική ψηφοφορία για το ψήφισμα. Άρχισε ψηφοφορία. Πέρασε. 17 προς 4 με 6 εποχές εγκρίνεται συγχαρητήρια στον εισηγητή, τον συνάδελφο Φιέλνερ. Και ερχόμαστε στο 19. Nein, also, liebe, liebe Kollegen. Συναδελφοί, σήμερα συνεδριάζουμε μέχρι τις και θα ψηφίσουμε μέχρι τις 6.30. Όχι παραπάνω, αλλά ούτε και πιο πριν. Και ό,τι μείνει αύριο το πρωί. Σημείο 19. Ρόμπερτ, η έκθεσή σου. Φαντάζομαι θέλεις να υπερψηφιστεί. Τροπολογίες στο σχέδιο προφορικής ερώτησης. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Απερίφθη. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά. Final vote on the draft resolution is amended. Αυτή τη φράση. Πέρας. Αυτό εγκρίνεται. Με μία αποχή. 15-11 μία αποχή. Και ερχόμαστε στο ψήφισμα. Συμβαστική τρία. Ηλεκτρονικά. πέρας. Εγκρίθηκε. 20 ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. 21 ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. 22 ηλεκτρονικά. Πέρας. Ενεκρίθη. 23 ηλεκτρονικά. Πέρασε. Απερίφθη. 24 ηλεκτρονικά. Πέρασε ενεκρίθη. 25 ηλεκτρονικά πέρασε απερίφθη Ρόμπερτ Παρακαλώ προφορική τροπολογία να κάνουμε χωριστή ψηφοφορία στην 26. Πρόεδρος. Μάλιστα. Χωρίς το πρώτο τμήμα. Ηλεκτρονικά. Πέρασε. Ενεκρίθη. Δεύτερο τμήμα. Ηλεκτρονικά. Πέρασε. Απορρίπτεται. 28. ηλεκτρονικά πέρας απερίφθη 29 ηλεκτρονικά. Πέρασε. Απερίφθη 30 ηλεκτρονικά. πέρασε απερίφθη. 31 ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. Τριάντα τρία. Ηλεκτρονικά. Πέρασε. Εγκρίνεται. 34. Ηλεκτρονικά. Πέρασε. Απερίθη. 35. Ηλεκτρονικά. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω πληροφορηθείτε ότι, ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε και την τροπολογία. Μετά την τροπολογία 31 πρέπει να ψηφιστεί και 32. Πρόεδρος, εμένα εδώ καταπίπτει αν ψηφιστεί η 31. Έχετε δίκιο όμως αυτό που είπατε, μου λέει η γραμματεία. Εγώ έχω μπροστά μου την, τη δική μου σειρά ψηφοφοριών. Παρακαλώ, ας ψηφίσουμε την 32 ηλεκτρονικά. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τριάντα πέντε. Ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. Τριάντα έξι. Προφορική. Αντιρρήσεις. Όχι. Ψηφίζουμε. Ηλεκτρονικά. Πέρασε. Εγκρίθηκε. 37. Έναρξη. Και λήξη. Εγκρίθηκε. Ρόμπερτ. Πληροφορική τροπολογία. για να είμαστε συνεπείς θα πρέπει να εφαρμόσουμε την τροπολογία που ανάφερα και στην αρχή. Πρέπει να ισχύσει το ίδιο. Αν δεν υπάρχει αντίρρηση φυσικά. Ερωτώ, στην προφορική αυτή τροπολογία υπάρχει αντίρρηση. Καμία. Τι ψηφίζουμε την 10 ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίθηκε. 40 ηλεκτρονικά. Επέρασε. Απορρίβεται. 42 ηλεκτρονικά. Πέρασε. Απορρίβεται. 43. Έναρξη. Πέρασε. απερίφθη συμβαστική 5 ηλεκτρονικά πέρασε απερίφθη 47 ηλεκτρονικά Πέρασε. Απερίφθη. 48. Ρόμπερτ. Μάλιστα, χωριστή ψηφοφορία για τη 48. Πρώτο τμήμα. Ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα. Ηλεκτρονικά. Πέρας. Απερίφθη. 49. Ηλεκτρονικά. Πέρασε. Απερίφθη. Συμβαστική 6. Ηλεκτρονικά. Πέρας εγκρίνεται. Συμβαστική 7 ηλεκτρονικά. Πέρας εγκρίθηκε. 57 ηλεκτρονικά. Πέρας εγκρίνεται. 58 δύο τμήματα. Το πρώτο, ηλεκτρονικά. Πέρασε. Απορρίπτεται. Το δεύτερο. Ηλεκτρονικά. Πέρασε. Απορρίπτεται. 59 ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. 60 ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίψετε. 63. Ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίψετε. 64. Ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. 65 ηλεκτρονικά πέρας εγκρίνεται. Εξήντα οχτώ ηλεκτρονικά πέρας απορρίπτεται. Συμβαστική 4. Ηλεκτρονικά. Πέρασε. Απορρίπτεται. 70. Ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. 71. Ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. 72 και 73 ταυτόσημες ηλεκτρονικά. πέρας απορρίπτεται 74 ηλεκτρονικά πέρας απορρίπτεται συμβαστική εννέα. ηλεκτρονικά πέρας Εβδομήντα οχτώ ηλεκτρονικά. Πέρασε. Εγκρίθηκε. 81 ηλεκτρονικά. Πέρασε. Απορρίπτεται. 82 ηλεκτρονικά. Πέρασε. Εγκρίνεται. Προφορική αντίρρηση. Μία αντίρρηση, Πρόεδρε. Αυτή η τροπολογία κατατέθηκε ως προφορική τροπολογία, αλλά καλύπτεται από άλλες τροπολογίες. Ρωτάω αν διαφωνείτε. Πέστε μου ναι ή όχι. Μου αρκεί. Ωραία. Κατέπεσε. Αιτιολογική σκέψη. Ένα ηλεκτρονικά. Πέρασε. Εγκρίνεται. Δύο. Ηλεκτρονικά. Πέρασε απορρίπτεται. Τρία, ηλεκτρονικά. Πέρασε. Απορρίπτεται. Συμβασική παραθμόν Ηλεκτρονικά. Πέρας Απορρίπτεται. έξι Χωριστή ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα. Ηλεκτρονικά. πέρας Εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα. Ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. Δύο. Συμβαστική. Ηλεκτρονικά. Πέρασε. Εγκρίνεται. Δέκα ηλεκτρονικά. Πέρασε. Απερίφθη. Έντεκα ηλεκτρονικά. Πέρασε. εγκρίνεται 12 ηλεκτρονικά πέρας εγκρίνεται 13 ηλεκτρονικά πέρας απερίφθη. 14 ηλεκτρονικά. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τελική ψήφος. Ηλεκτρονικά. Πέρασε. Ναι, εγκρίνεται με 17, 10 και μία αποχή. Συγχαρητήρια στο ραμπέτσι Περνάμε τώρα στο σημείο 20 της ημερησίας διάταξης. Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Κοινότητας της Ανατολικής Αφρικής. Έχουμε εδώ την... το σχέδιο Ευρωπαϊκής Ερώτηση. Ψηφίζουμε μπλοκ καταρχήν όλων των ομάδων. Άρχισε ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 1. Και αυτή στο μπλοκ. Ωραία. Άρχισε ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Άρχεται. Πέρα. Εγκρίνεται. Και τώρα, τελική ψηφοφορία. Άρχισε η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια, Χέλμουτ. Ε, το είπα στον εαυτό μου. Και περνάμε στο σχέδιο ψηφίσματος. Ψηφίζουμε μπλοκ όλων των ομάδων. άρχιψη ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 16. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 43. Σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα την ψηφοφορία. Πέρας. γίνεται δεύτερο τμήμα. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεκαεφτά. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. για 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 20. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Ναι, μία ψήφο. Ψήφο ψηφία. Τροπολογία 21 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Όσο πάει και λιγοστεύουμε εδώ. Τροπολογία 22, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία παριθμών 1. Διαφωνεί κανένας. Όχι. Ψηφίζουμε. Άχι ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 23. Άκρη ψηφοφορία. Πένας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχισε ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Άρχισε ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Άρχισε ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 27. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 28. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 29. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία παριθμών 3. Διαφωνίες. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 30. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 31. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 32. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 33. Άρχη ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 34 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Ευτυχώ που ήταν, δεν ήταν εδώ ο Κρίστοφερ να ακούσει τι ελέγχθη εδώ. 35 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 36. Άρχισε φοφορία. φοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 37. Άρχεται. 37 λέω, ναι. Πέρας. Απορρίπτεται. 38. Άρχεται. Πέρας. Πονά τα δάχτυλά σου πάτα στην κάρτα συνεχώς. Απορρίπτεται. 38. Άρχεται. 39, συγγνώμη λέει ο πρόεδρο. Πέρα. 39. Εγκρίνεται. 40. Άρχεται. Πέρα. Εγκρίνεται. 41. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 42. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 47. Άρχη φοβορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 48. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 49. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 51. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 53. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 54. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 56. Άρχεται. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, 55. Ναι, ναι, ναι, 55. Λοιπόν, τροπολογία 55, η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 56. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 57. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 58. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 59. Άρχεται. Πέρας. Το Τροπολογία 61. Άρχεται. Και εγώ λέω, πρόεδρος θα το σχολείο ήταν εκτός μικροφόνου. Πέρας ψηφοφορίας. Απερίφθη. Τροπολογία 24. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. δύο καταπίπτει. Φτάνουμε στην Στην τροπολογία λέω. Δεν είμαι τόσο βληγορό. Λοιπόν, φτάνουμε στην 63. Ναι, στην 63. Άρχισε η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για την 63. Πέρασε τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 70. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 71. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 72. Άρχιψη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 73. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 74. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 75. Άρχεται. Η 74 απερίφθη, γι' αυτό πρέπει να ψηφίσουμε 75. Λοιπόν, πέρασε ψηφοφορία για 75. Εγκρίνεται. Και καταπίπτει 76, 77 και 87. Και πάμε στην τροπολογία 78. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 79. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 80. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 81. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία παριθμών 2. Διαφωνεί κανένας? Όχι. Ψηφίζουμε. Την πληροφορική τροπολογία αυτή. Άρχεται. Ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 84. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στη βασική τροπολογία υπαριθμών 1. Άρχισε ψηφοφορία. Ρόμπερτ, το ερώτημα είναι για σένα, από είναι συνάδελφο Φόρτ. Θέλεις να ζητήσεις την ίδια προφορική τροπολογία. Ναι. Ναι. Προφορική τροπολογία να είμαι ευθυγραμμισμένος με το υπόλοιπο. Ωραία. Ψηφίζουμε, αν δεν διαφωνεί κανένας με την προφορική τροπολογία. Την συμβαστική τροπολογία παριθμών 1, όπως τροποποιήθηκε προφορικά. Άρχινη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμφωνήσατε, νομίζω υπερψηφίσατε για να καταπέσουν τόσα πολλά εδώ, ε. Να προχωρήσουμε γλίγορα. 102. Το 102. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Το Τροπολογία 105. Άρχεται η ψηφοφορία. Όχι. 105 λέω. Ναι. Πέρασε ναι. ε, ψηφοφορία. Δεν κρίνεται. 95. Άρχισε ψηφοφορία. 95 λέω. Πέρασε ψηφοφορία. Απερίφθη. Τροπολογία 99. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. 101. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απερίφθη. Τροπολογία 106. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 107. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 1. Πέρας. Εγκρίνεται. 2. Άρχιε ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τρία. Άρχιψη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία τέσσερα. Άρχιε ψηφοφορία. Geschlossen. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 6. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 7. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 8. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 9. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 10. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 11. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 14. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. 16 υπέρ, 9 κατά και καμία αποχή. Ωραία. Κλείσαμε και το σημείο αυτό της μερικής διάταξης, το 20, και περνάμε στο σημείο 21. Λοιπόν, υπάρχει παράκληση να κάνουμε μια σύντομη διακοπή. Καταλαβαίνω ορισμένοι έχουν κάποιε ανθρώπινε ανάγκες. Τρία-τέσσερα λεπτά, ένα σύντομο διάλειμμα. Εντάξει. Ευχαριστώ.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 Ωραία λοιπόν ε, καθίστε και πάμε στην έκθεση του συνάδελφου, του συνάδελφου Κασπάρη. Λοιπόν, προφορική, σχέδιο προφορικής ερώτησης. Έπεσαν καλύτερα να δουλεύουμε τώρα με ανάτες της χειρός. Πρόεδρος. Ωραία, ας το δοκιμάσουμε. Για να δούμε πώ τυχόν πάει καλύτερα. Λοιπόν, τροπολογία 1 και 4, αμπλοκ. Υπέρ. Κατά. Απολύτω. Τροπολογία 2 υπέρ κατά Απορρίπτε. τροπολογία 3 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές Απορρίπτε. δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές Απορρίπτε. 5 υπέρ κατά εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τελική ψηφοφορία με ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται με 22-1-1. σχέδιο ψηφίσματος. Αμπλοκ. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογίες 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 26-27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται προφορική 3 αντίρρηση όχι. Ναι. Also, äh, wir sind jetzt beim Nummer 3. Wer ist dafür? Τροπολογία του 3. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην προφορική τροπολογία 29. Υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 30 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 34 καταπίπτει. 35 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 36 προφορική τροπολογία διαφωνεί κάποιος όχι ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 38 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε αυτό καλύτερα. Την 40 να ελέγξουμε παρακαλώ. Άρχισε ψηφοφορία. Πέρας. 10 υπέρ, 15 κατά. Ναι. Απορρίπτεται. Τροπολογία 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 43 και 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 47 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 81 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχέ, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχέ, απορρίπτεται. Τροπολογία 49 υπέρ. Κατά αποχέ, εγκρίνεται. 50 και 51 υπέρ. Κατά απόχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 52 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 53 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Εγκρίνεται, ναι, ναι, εγκρίνεται. 54 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία υπαριθμών 1. Διαφωνεί κανένας, όχι, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. πέπτη, τροπολογία 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 2 υπάρχει μια διαφωνία. Όχι, ωραία. Ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια ψηλά να σα βλέπω. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Που ερνάμε τώρα στην συμβαστική τροπολογία 1. Υποθέτω ότι και εδώ ισχύει αυτή η προφορική τροπολογία, Ρόμπερτ. Ωραία. Όπω έχει τροποποιηθεί, συμφωνούμε Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Θα καταπίπτει αυτό ή τούτο. Και φτάνουμε στην 69. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ναι, ναι, ναι, εντάξει. εντάξει. Τροπολογία 71, ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία ε, ηλεκτρονικά για την 71. Πέρας. 11 υπέρ 15 κατά. Σωστά το είδα. Τροπολογία 72 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία καταπίπτουνε 77. 77 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3. 78 να ελέγξουμε. Ευχαρίστω. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για την 78. Πέρας. Ναι, 16 υπέρ 10 κατά. Σωστά. Είναι κρίθη. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 3. Ναι, σωστά το είδα. Α, λοιπόν, 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 82, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 87 υπέρ κατά Απορρίπτεται. Τροπολογία 88. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 89. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 92. Υπέρ. Κατά. Για να το ελέγξουμε αυτό καλύτερα. Για την 92 ηλεκτρονικό έλεγχο παρακαλώ. Πέραση ψηφοφορία. 12 προς 14. Απερίφθη. Περνάμε στην τροπολογία 93. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η ίδια πλειοψηφία. Απερίφθη. 94. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 95. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 97 υπέρ κατά αποχές για να το ελέγξουμε καλύτερα την 97 παρακαλώ ηλεκτρονικός έλεγχος για την 97 Άρχιψη ψηφοφορία πέρας 11 υπέρ, 15 κατά. Απορρίπτεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 100 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 104 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 105 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 109. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 110 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 113 προφορική τροπολογία διαφωνεί κανένας όχι ωραία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά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 Ένα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Φτάνουμε τώρα στην τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά βέβαια άρχη ψηφοφορία πέραση ψηφοφορία. 16 ψήφοι υπέρ και 7, 2 κατά και 7 αποχές εγκρίνεται Μπορούμε να συγχαρούμε τον κύριο Κασπαρή. Όπω είναι ικανοποιημένο νομίζω με το αποτέλεσμα. Και φτάνουμε, θα τα καταφέρουμε, δεν θα το φανταζόμουν ποτέ. Αν, αν, είχα κάνει, αν είχα βάλει στοίχημα, θα είχα χάσει σίγουρα. Ε. Δεν το φανταζόμουν ποτέ. Λοιπόν, φτάνουμε τώρα στο σημείο 22 τη ημερησία διάταξη. Ε, προ... Σχέδιο προφορική ερώτηση καταρχήν. Έχουμε μια προφορική τροπολογία. Διαφωνεί κανένα. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Για να το ελέγξουμε καλύτερα. Δεύτερο τμήμα της προφορικής τροπολογίας υπεριθμών 1. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. 11 υπέρ 15 κατά. Απερίφθη λοιπόν. Προφορική τροπολογία περίπου 2. Υπάρχει διαφωνία? Όχι. Ποιος είναι υπέρ? Κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία για την ε, προφορική ερώτηση. Ποιος είναι υπέρ? Α, ηλεκτρονικά καλύτερα. Λοιπόν, ηλεκτρονικά. Άρχη ψηφοφορία. Τελική ψηφοφορία. Πέρας. 25 υπέρ, ε, μία ψήφος κατά. Και περνάμε τώρα στην... Για να δω. Στο σχέδιο ψηφίσματος και περνάμε με την... καταρχήν με ψηφοφορία on block. Ποιος είναι υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. Τροπολίγια 14, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές να σηκώνετε τα χέρια σας παρακαλώ 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αλλά δεν το βλέπω, να σηκώνετε τα χέρια σας. Συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία περιθμών 1. Διαφωνεί κανένα. Όχι. Λίγη ησυχία παρακαλώ. Θα τα καταφέρουμε. Υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25. Υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. Αγαπητοί συνάδελφοι. Αρίφ και Καρνέλα, σας παρακαλώ. Τροπολογία 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Για να το ελέγξουμε αυτό ηλεκτρονικά. Για την 26 παρακαλώ. Άρχεται. Πέρας. 15 υπέρ, 11 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν. 27 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 31 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία υπαριθμών 2. Υπάρχουν διαφωνίες. Α, καταπίπτει, καταπίπτει. Ναι, ναι, ναι. Τροπολογία 32. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 33. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ Κα... υπέρ λέω 34 κατά αποχές εγκρίνεται Ναι, παραλάβουμε. Ήταν σοβιάστηκα πάρα πολύ. Τροπολογία 34. Ποιος είναι υπέρ της 34 παρακαλώ. Μα ψηφίσαμε 33. Γιατί έχουμε βάλει εδώ. Λοιπόν, να επαναλάβουμε την 33. Ίσως βιάστηκα πολύ. Επαναλαμβάνουμε την 33. Ποιος είναι υπέρ της 33 παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 36 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 40 υπέρ. Κατά Αποχές απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Για να το ελέγξουμε. Για τη 41 ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Πέρας πληροφορίες. 14 υπέρ, 11 κατά. Ναι, εγκρίνεται. Τροπολογία 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 μπλοκ 49 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία. Α, καταπίπτει. Καταπίπτει. Ωραία. 50 και 51. Επίσης, 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 53. Υπέρ. Κατά. Για να ελέγξουμε. Για την 53 παρακαλώ. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας πληροφορίες, Απερίφθη 2 προς 16 με 8 αποχές. Η 54 σε δύο τμήματα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτει δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίπτεται. Η 56. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 57 υπέρ κατά αποχές για να το ελέγξουμε την 57 να ελέγξουμε Άρχιτη ψηφοφορία πέρας 11 υπέρ 14 κατά απερίφθη τροπολογία 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται βασική τροπολογία περίπτωση 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 60 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 62 υπέρ. Κατά αποχές μάλλον απερίφθη. Τώρα Να ελέγξουμε. Να ελέγξουμε. Την 62 παρακαλώ. Άρχιε ψηφοφορία. Πέρας. Ναι, ναι, απερίφθη. Και περνάμε στην τροπολογία 64, υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται και καταπίπτει 68 και περνάμε στην συμβαστική τροπολογία υπεριθμών 5. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 69 υπέρ κατά αποχές μάλλον απερίφθηκε αυτό 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 6 με την προφορική τροπολογία πάντα που είχαμε παν μέχρι στιγμή. Δεν διαφωνεί κανένα για την προφορική τροπολογία. Ωραία, ψηφίζουμε τη συμβαστική υπαριθμών 6. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε στην τροπολογία υπαριθμών 71. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και πάμε τώρα στη συμβαστική τροπολογία παριθμών 7. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στην 79. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 81. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 83. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική τροπολογία υπερθυμών 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Να σηκώνετε τα χέρια σας παρακαλώ, τελειώνουμε. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πολύ ωραία, πολύ ωραία έτσι. Τροπολογία 7 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 σε δύο τμήματα. Υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται νομίζω. Και φτάνουμε στην... Φτάνουμε λέω στην τελική ψηφοφορία. Και έχει ζητηθεί ονομαστική, ονομαστική ψηφοφορία από τον Γκλινφόρτ. Και αυτό θα κάνουμε τώρα. Άρχιτη ψηφοφορία. Δεν θέλουμε να έχουμε μακρύ τώρα. Πέρας. 23 ψήφοι υπέρ, 2 ψήφοι κασά. Τελειώσαμε αυτή τη μακρά ψηφοφορία. Ευχαριστώ όλους όσοι συμμετείχαν, ευχαριστώ τους διερμηνείς. Σας εύχομαι καλό βράδυ και αύριο, αύριο δεν έχουμε συνεδρία στις επιτροπές μας. Τελειώσαμε. Και ευχαριστώ τους διερμηνείς για